Κληρωθεί η πρώτη ανάγνωση. Σημείο 3. Ή μάλλον σημείο 4. Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων. 19 και 20 Νοεμβρίου του 2018. συμφωνείτε όλα αυτά καταπληκτικά πρακτικά. Αν ναι, οπότε θα περάσουμε στο σημείο 5. Να καλωσορίσω την ε, κυρία Μαρία Κοτσέβα, Γενική Διευθύντρια της Eurostat. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Θα σας δώσουμε και το λόγο για 10 λεπτά να μας κάνετε μία εισαγωγική παρέμβαση και έπειτα θα έχουμε ερωταπαντήσεις, πολλές ε, για πέντε λεπτά. Δεν είμαστε και πολύ σήμερα. Οπότε μπορούμε να παρατείνουμε το χρόνο για τον καθένα σε περισσότερα από πέντε λεπτά και εσείς δεν έχετε αντίρρηση. Η σημερινή συνεδρίαση γίνεται με βάση τον κανονισμό 223 του 2009 που λέγεται ότι η Γενική Διευθυντήρια, ο Γενικός Διευθυντής ε, κατά περίπτωση θα είναι αρμόδιος για τις αρτιστικές δραστηριότητες και θα παρουσιαστεί, θα παρουσιάζεται τέλος πάντων στις αρμόδιες επιτροπές, την ΕΚΟ δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, για να συζητά ζητήματα που απτούνται τη στατιστική διακυβέρνηση μεθοδολογίας και στατιστικής καινοτομίας. Και η κυρία Κοτσέβα ακριβώ για αυτό το λόγο βρίσκεται εδώ και τη δίνω αμέσω το λόγο και την ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη και που δεν έχουμε σημαντική προσέλευση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλου σα. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Ενώπιόν σας πριν από ένα περίπου χρόνο ήρθα όταν ορίστηκα νέα διευθύντρια. Και ήταν ιδιαίτερα καρποφόρη χρονιά αυτή όσον αφορά τη συνεργασία μας. Θεωρώ λοιπόν πάντα την συνεργασία και αυτή την ανταλλαγή απόψεων όπως είναι η σημερινή κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που βοηθάει επίσης να προωθήσουμε και τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα με τον κύριο Γκουλτιέρ είχαμε συμφωνήσει ότι θα σας παρουσιάσουμε μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια που έχω πει και άλλες φορές, δεν θα σας φορτώσω με τεχνικές λεπτομέρειες, θα τις συνοψίσω όμως ως εξής. Μετά από την πρώτη φορά που παρουσιάστηκα εδώ ενώπιόν σας, ένα χρόνο μετά, είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε συνεργασία με τις χώρες μέλη σε τρεις τομείς. Πρώτον, στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ε, στατιστικών δεδομένων. Δεύτερον, να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την ψηφιακή τεχνολογία και τις νέες πηγές δεδομένων, ώστε να είναι ε, περισσότερο κατάλληλη και με περισσότερες λεπτομέρειες η παραγωγή στατιστικών δεδομένων μας. Και η τρίτη πτυχή είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία και η διάδοση των στατιστικών δεδομένων. Τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στο input. Θέλω όμως να επικεντρωθώ στο εξή. Είμαι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαιρετική δουλειά που κάνουμε σε διάφορους κανονισμούς στο πλαίσιο τα τελευταία χρόνια στα στατιστικά όσον αφορά τη γεωργία, τα κοινωνικά δεδομένα, τα στατιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων, τη μετανάστευση. Οι φάκελοι βρίσκονται φυσικά σε διαφορετικό επίπεδο ο καθένας, αλλά δεν υπερβάλλω για το ότι χάρη στην συμμετοχή των συναδέρφων σας στους τριμερείς διαλόγους ε, καταφέραμε να καταρτήσουμε τη γραμμή μας όσον αφορά το μέλλον των επίσημων στατιστικών δεδομένων στην Ευρώπη. Και θα σας δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Εμείς, ακόμα και με καινοτόμα εργαλεία, με πιλωτικές μελέτες, ε, ε, μελέτες σκοπιμότητας ε, κλπ. Φροντίζουμε για την διάδοση των στατιστικών δεδομένων και καινοτομήσαμε θέτοντας το πλαίσιο της ρύθμισης, αλλά φροντίζοντας να ανταποκριθούμε και σε νέα αιτήματα στο κατάλληλο πάντα επίπεδο. Και επίσης στην νομοθεσία χρησιμοποίησαμε την ευκαιρία να συμπεριλάβουμε νέα τεχνολογία, νέες τεχνολογίες, ε, διοικητικές λύσεις, αλλά και κάποιους μηχανισμούς, κάποια εργαλεία, όπως αυτά που κυκλοφορούν εδώ πολύ. Ελπίζουμε σε αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κλείσουν όλοι οι φάκελοι. Να ξέρετε ότι θα είμαι πάρα πολύ ευτυχής ως Γενική Διευθύντρια γιατί έτσι μετά θα περάσουμε και εμείς τη κατεξοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την επικοινωνία. Πέρυσι, όταν συναντηθήκαμε, σας είπα ότι δεν είχα πια την πολυτέλεια να είμαστε η μόνη πηγή στατιστικών δεδομένων και ότι υπάρχει ψηφιακή διασύνδεση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλές πηγές. Διερευνήσαμε λοιπόν προκειμένου η ιστοσελίδα μας να γίνει περισσότερο φιλική προς το χρήστη. Επικεντρώσαμε την προσοχή μας στους πολίτες, στα πράγματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους. Συμπεριλάβαμε διαδραστικά εργαλεία με διάφορες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης και να επεκταθεί περισσότερο στην έρευνά του. Ερευνήσαμε επίση και οπτικά τι μπορούμε να κάνουμε στην ιστοσελίδα μας με διαγράμματα, δηλαδή τα δεδομένα μας, ναι, διαδίδονται, αλλά και η ζωή συνεχίζεται. Οπότε και οι χρήστες και εσείς να μπορείτε συνεχώς να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα μας για να λάβετε και τις αποφάσεις που καλείστε να λάβετε. Επίσης, αρχίσαμε και συζητήσεις με τους fact-checkers Δίνουμε δηλαδή τα δεδομένα μας και αρχίσαμε να υπογραμμίσουμε περισσότερο και το θέμα ε, της δυνατότητας κατανόησης των στατιστικών δεδομένων από τον κόσμο. Ε, υπήρξαν κάποιες δράσεις τις οποίες συμμετείχαν πολλές χιλιάδες νέοι. Είναι και αυτός ένας τρόπος για να προωθήσουμε το έργο μας στο μέλλον. Πολλά μένουν βέβαια ακόμα να γίνουν και μια που και εσείς φτάνετε στο τέλος της δικιάς σας θητείας, ελπίζω οι άνθρωποι που θα σας ε, διαδεχθούν θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα επίσημα στατιστικά δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Και θα τελειώσω με ένα παράδειγμα από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να βρίσκουμε αλγορίθμους και να τους χρησιμοποιούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά το να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα ε, στις, στην παραγωγή στατιστικών δεδομένων ε, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντε ρόλο. Η ηθική, το τι μπορεί, τι πρέπει, τι δεν πρέπει να κάνει κανείς. Οπότε αυτή η συνεργασία μεταξύ μας ελπίζω να συνεχιστεί και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέω, για την εισαγωγή αυτή. Ξεκινάει η συζήτηση. Από το ΕΛΚ δεν βλέπω κανέναν εδώ, άρα θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στη συντονίστρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Περβάν Μπερέ. Ευχαριστώ. πολύ. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο έχει περάσει από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σα και είσαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάλι. Χαιρετίζω τον ορισμό σας και βλέπω ότι δικαιολογείται απόλυτα. Δεν έχω πολλές ερωτήσεις. Μάλλον έχω πολλές ερωτήσεις και θα μία-μία θα τις κάνω. Κάτι γενικό πρώτα απ' όλα, το οποίο είναι κάτι που μας απασχολεί εμάς πολιτικά. Ποιες είναι οι συνθήκες που απαιτείτε εσείς από τις χώρες μέλη, τι πληροφορίες απαιτείτε και πώς εσείς ε, διαπιστώνεται κατά πόσο έχουν υλοποιήσει τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που μας απασχολεί. Εμένα με ενδιαφέρει να έχουμε έναν πίνακα κάπως παράλληλο για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον προπολογισμό των χωρών ε, μελών. Όλα αυτά βέβαια πέρασαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι παλιά ιστορία. Αλλά το αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι η υλοποίηση των 17 στόχων. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν δεν έχουμε τα δεδομένα ε, που να είναι κοινά, αν δεν έχουμε κοινού ορισμούς για το τι καλύπτουμε, δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε μια πολιτική στρατηγική. Οπότε τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό, τι έχει γίνει, τι ετοιμάζετε, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας τι περιμένετε από τις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπερέσα. Για λόγους αποτελεσματικότητας λέτε πώς μπορούμε να θέτουμε τα ερωτήματα. Πράγματι, συμφωνώ ότι δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία για τη Eurostat. Έχουμε τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Είναι θέμα και πολιτικής βούλησης, πολιτικής δέσμευσης και απόφασης. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή θα καταβάλει προσπάθεια την επίτευξη των στόχων αυτών που υπερβαίνουν το πεδίο των στατιστικών. Δεν είναι στατιστική υπόθεση. Τα τελευταία δύο χρόνια καταρτήσαμε νομίζω πριν δύο χρόνια την πρώτη έκθεση, έλα έληφθη απόφαση οι πολιτικές που εφαρμόζουν προτεραιότητες της Ένωσης και διάφορες πολιτικές κομισιών συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και εμείς είχαμε ως να καταθέσουμε προτάσεις για δείκτες που ε, ε, βοηθούν στην εκπλήρωση. Αλλά δεν ήταν εύκολο με το 2020, την Ευρώπη 2020 που είχαμε κάποιους ε, στόχους απομοντήμους και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δείκτες. Με βάση τη στατιστική μας γνώση και τις συζητήσεις με διάφορους εμπλικομένους φορείς και με την Κομισιόν, με τις ΜΚΟ, με τα κράτη-μέλη, η Eurostat κατάρτισε τις προτάσεις της και εκπώνησε μια έκθεση που δίνει ουσιαστικά τη στατιστική εικόνα, πώς έχει κατάσταση, πού βρισκόμαστε, ε, απέναντι στους στόχους αυτούς ε, των Εθνών και η ιδέα μας ήταν να δώσουμε στο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες με διδραστικό τρόπο. Αναθεωρήσαμε για μια ακόμη φορά τη δέσμη δικτών στα τέλη του προηγούμενου έτους και η επόμενη έκδοση θα είναι έτοιμη τον Ιούλιο του 2019. Έτοιμη για το πολιτικό φόρουμ ψηλού επίπεδου σε επίπεδο ΙΕ. Οπότε και θα συζητηθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξη. Έτσι έχει κατάσταση. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο αυτό που σα είπα. Πρόεδρος. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ο Βόλφ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Να σας συγχαρώ που αναλάβατε το πολύ σημαντικό αυτό καθήκον. Η Eurostat ε, πολλές φορές υποτιμάται ε, η σημασία δηλαδή αυτού του οργανισμού υποτιμάται. Και πρέπει να πω ότι για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κατ' εμεύρο η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία έχει να επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. και η πρώτη μου ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, είστε πραγματικά ικανοποιημένοι. Γνωρίζουμε ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν κάποια προβλήματα γιατί οι εθνικέ στατιστικέ υπηρεσίε ε, δεν επεδείκνυαν το δέον πνεύμα συνεργασία. Και το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Ο τέο ε, διευθυντής της ελληνικής ε, εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, ο κύριο Γεωργίου, από την κυβέρνηση μέχρι και δίκη παρεπέμφθη δίκη για ψευδή στοιχεία ε, και παραποίηση στοιχείων. Το μόνο όμως που έκανε ουσιαστικά ήταν να αναζητήσει τα ε, σφάλματα των προκατόχων ε, του προκατόχου, να τα διορθώσει και να διαβεβαιώσει ότι από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η υπηρεσία του θα είχε πλέον θα έδινε τα σωστά στοιχεία. Προσπαθείτε εσείς να έρθει σε αισιοπέραση η υπόθεση αυτή. Διότι όπως γνωρίζουμε δεν βλάπτει αυτή η υπόθεση μόνο την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και την κυβέρνηση βέβαια, αλλά είναι και ένα τεράστιο ε, πρόβλημα ε, προσωπικό, ανθρώπινο, για τον άνθρωπο αυτό που χρειάστηκε να επενδύσει και πάρα πολλά ε, κονδύλια και δεν μπορεί να είναι στην πατρίδα του γιατί κινδυνεύουν να τον συλλάβουν ε, ε, αμέσως. Είμαστε μία ένωση δικαίου. Εδώ βλέπουμε πραγματικά μεγάλη παραβίαση της νομοθεσίας σε αυτή την περίπτωση από την κυβέρνηση τότε. Και πραγματικά θέλω να μου πείτε εσείς τι κάνετε για να δοθεί ένα έσω πέρα σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ που αντιλαμβάνεστε και εκτιμάτε το ρόλο της Eurostat. Σύντομα να πω ότι ναι, είμαι ικανοποιημένη από τη συνεργασία με τα κρατημέλη στην επίσημη στατιστική. Η επίσημη στατιστική, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη ζωή. Και όταν αλλάζει η ζωή και έχουμε νέες προκλήσεις και νέες απαιτήσει, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Αν υπάρχουν λοιπόν ζητήματα, θα πρέπει να δούμε από κοινού ε, τι, πώς επηρεάζονται την ζήτηση επίσημων στατιστικών. Και δεν είναι εύκολα όλα τα θέματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, τι στατιστικέ έρευνε που θα οργανωθούν την επόμενη εξαετία για να σα δώσουμε πληροφορίε. Τι πληροφορίε πρέπει να σα τι δώσουμε αύριο. Αυτέ είναι οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε και αυτά τα μέσα και τα νομικά μέσα μεταξύ άλλων με τα οποία θα βοηθήσουμε ε, να οργανώσουμε την απόκρισή μα ε, για το μέλλον. Για την Ελλάδα, ε, καταρχά να πω δύο πράγματα. Η Eurostat, ε, όποια ευκαιρία είχε, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκανε, την έχουμε αξιοποιήσει για να επαναλάβουμε και να ξαναεπαναλάβουμε ότι από το 2010 η Eurostat ποτέ δεν είχε κάποια επιφύλαξη για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει επικυρώσει τα δεδομένα. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία από το 10 και μετά για τα δεδομένα. Εμεί όμω ε, τρέφουμε κάθε σεβασμό στο νομικό σύστημα στην Ελλάδα και δεν παρεμβαίνουμε στη δικαστική διαδικασία. Παρακολουθούμε την όλη δίκη με ανησυχία Υπήρξαν ε, συγκεκριμένα βήματα τα οποία ε, έγιναν τα τελευταία χρόνια ώστε στο νομικό πλαίσιο να εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε εκ νέου αντίστοιχες περιπτώσεις. Ένα δεύτερο πολύ συγκεκριμένο ε, θέμα, ένα κόστος, identification cost που μπήκε το 2016 και ήταν ένας τρόπος για την αποζημίωση του κυρίου Γεωργίου. Ο αντιπρόεδρο των ο Πρίστροπο ε, και η Μαριάν Τάισεν, ενώ δεν ήταν η Eurostat μόνο, που εξέφρασαν πολύ ξεκάθαρε κατηγορηματικέ απόψει. Εμεί ω Eurostat συνεχίζουμε και επιβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα είναι ποιοτικά από την Ελλάδα και αξιόπιστα. Να δώσω ξανά το λόγο στην Περβάς Μπερέσσα, Παρακαλώ, Περβάς. Ευχαριστώ πολύ. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με τη συλλογή πληροφοριών για δημοσιονομικά θέματα. Καθότι, όπως γνωρίζετε, τα κράτη-μέλη, βάση οδηγίας, πρέπει να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για για τα φορολογικά και τις ε, διευθετήσεις που προβλέπουν. Ε, εδώ λοιπόν ε, θα ήθελα να μου πείτε τι κάνετε με τη συλλογή αυτών των δεδομένων Και δεν είναι αυτή καθεαυτή φόρο διαφυγή αυτή. Είναι όμως νομοθεσία που προβλέπουν τα κράτη-μέλη και στην ουσία κάπως αποστραγγίζει το δημοσιονομικό τους εισόδημα. Είναι κάτι λοιπόν που μας ταλανίζει αυτό και είναι δύσκολο να βρούμε απάντηση ποιο είναι ο πραγματικό συντελεστή φορολόγηση των εταιρεών των εταιρεών διαφόρων κρατών μελών. Διότι ξέρετε ότι είναι σημαντικό και η δική σα η θετική προβολή να βελτιωθεί ω προς αυτό το θέμα. Θα έχω και άλλε ερωτήσει εάν δεν έρθουν άλλοι συνάδελφοι να κάνουν τι δικέ του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτήν την κέρια ερώτηση. Να ξεκινήσω από τη δεύτερη, διότι ναι, θέλουμε να προβάλλουμε τις στατιστικές μας συλλογέ και τα δεδομένα μας, ιδάλλως δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Η φορολογία και οι φορολογικοί συντελεστέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντικείμενο κοινή δημοσίευση με την ταξούτη, τη Γενική Διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνει στοιχεία και αναλύσει Και έτσι τα διαθέσαμε στους οικονομολόγους και όσους τα μελετούν τα θέματα αυτά για να τα αξιοποιήσουν. Ως προς το φορολογικό χάσμα, θα ξέρετε ότι το ε, περίφημο ΑΕΠ πρέπει να είναι διεξοδικό, να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και την άτυπη οικονομία Και δεν θα ήταν, νομίζω, υπερβολή να πω ότι είμαστε από τους πρωτοπόρους στον κόσμο στη συλλογή τέτοιων στοιχείων και ότι καταγράφουμε και τις δραστηριότητε ακόμα και τις παράνομες ε, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, διακίνηση ναρκωτικών, το εμπόριο οποιοδήποτε παράνομου προϊόντο. Ε, τα κράτη-μέλη πρέπει λοιπόν να τα μετράνε αυτά τα πράγματα και να τα περιλαμβάνουν στον ΑΕΠ στο ΕΠ. Όμως δεν έχουμε ακριβώς καταγράψει το φορολογικό χάσμα, δεν το έχουμε ως ξεχωριστό ποσοστό στο σύνολο του ΑΕΠ. Απλώς προσπαθούμε να καταγράψουμε όλες τις δραστηριότητε, ώστε συνολικά τα στοιχεία μας για το ακαθάριστο εθνικό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι σωστά. Ευχαριστώ. Επερώτηση στην ερώτηση της υπερβάνησης. Το θέμα της υποβολής εκθέσεων αναχώρα. Εδώ είναι μια περίπτωση όπου ήμασταν ε, ξεκάθαροι στο κοινοβούλιο τουλάχιστον και ιδίω η ομάδα μου πιστεύουμε ότι η υποβολή εκθέσεων αναχώρα είναι σημαντική, ιδίω εκεί που δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικέ. Τι φόρο πληρώνουν, για ποιο πράγμα και τι είναι απαραίτητο για να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε ώστε η νομοθεσία να είναι καλή και εντός των κρατών μελών, αλλά μετά και σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προ στιγμή το ντοσχέ αυτό δεν έχει προχωρήσει στο Συμβούλιο, έχει μπλοκαριστεί και δεν υπάρχει πλειοψηφία ώστε να είναι δημόσια τα στοιχεία της υποβολής εκθέσεων αναχώρα. Κατά την άποψή σας, ποιο θα ήταν ε, το ιδανικό, ε, πώς θα ήταν καλή κατάσταση για να έχουμε δημόσια υποβολή εκθέσεων αναχώρα. και πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα αποτελεσματικά από στατιστικής σκοπιάς. Τι πράγματα, τι χρειάζεστε ώστε η Eurostat να βοηθήσει εδώ. Να υπάρχει μια καλή συνολική εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Με το φόρο στις εταιρείε εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αυτό με επαναφέρει στην προηγούμενη ερώτηση. Δεν έχουμε προβλήματα με τα κράτη-μέλη Εάν λοιπόν καλά κατάλαβα, θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε λέτε στον αντίκτυπο των πολυεθνικών και τη δική του τη δραστηριοποίηση στι εκθέσει ένα χώρα. Διότι η αλυσίδα παραγωγή αξιών και εισοδήματο είναι, είναι κοινή για όλε τι χώρε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ποσά ε, μπορούν να κερδίζουν σε κάθε χώρα. Μικτά τουλάχιστον ε, και με τι νομικό καθεστώ λειτουργούν ω εταιρείε στην κάθε χώρα. Ε, το κοιτάζουμε λοιπόν αυτό για τι πολυεθνικέ. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα στατιστικά στοιχεία και τη ροή πληροφοριών σχετικά, αλλά χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών ε, πολυδιάστατη εδώ. Γι' αυτό το σχετικό πλαίσιο για τι εταιρικέ στατιστικέ είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι η κατάλληλη υποδομή για να επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων και μικροδεδομένων μεταξύ των χωρών. Ιδάλω είναι δύσκολο να απεικονίσουμε ε, το τι συμβαίνει σε κάθε λεπτομέρεια. Αλλά δεν υπόσχομαι ότι ο δρόμος θα είναι ομαλός και εύκολος. Είναι θέμα εθνικών αριθμών και είναι θέμα ανταλλαγής στοιχείων ώστε να προσθεθούν σε αυτά που έχει το κάθε κράτο μέλος και να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει ε, με τις ροές εκτός ε, των εταιριών και εκτός των χωρών ε, της κάθε χώρας όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Φυσικά αυτό είναι μέρος των φόρων επίσης. Έχετε ακόμα λίγα λεπτά. Είμαστε στη διαδικασία CatchDI. Τι άλλη ερώτηση. Υπερβάνω σε λίγο, θα ρωτήσει ακόμα κάτι, αλλά δώστε μου την ευκαιρία να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα. Η αναχώρα εκτός θα επιτρέψει στην Eurostat να καταλαβαίνει καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα. Αν δεν υπάρχει αυτή η δημόσια αναφορά, το μόνο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να έχετε ε, ανταλλαγή μόνο δεδομένων, κάτι το οποίο δεν προβλέπετε αυτό κάθε αυτό ακόμα. Οπότε, σωστά έχω καταλάβει ότι αν δεν υπάρχει public στην αναχώρα αναφορά, τότε η Eurostat δεν θα μπορέσει να καταλήξει σε καλύτερα δεδομένα. Απάντηση. Ναι. Αλλιώς όντως θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε άλλες πηγές αν δεν δημοσιοποιούνται τα δεδομένα από τις χώρες. Μην νομίζετε, δεν θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε άλλες πηγές, άλλους τρόπους. Ε, κύριε Μπερές, ε, ωραία, μια που μπορούμε να έχουμε διάλογο, θα συνεχίσω με αυτό το προνόμιο που μου δίνετε. Λοιπόν, η πρώτη μου επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το εξή. Από τα δεδομένα που συλλέγεται, ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται για τις κοινωνικές ανισότητες και μεταξύ χωρών αλλά και μέσα στην ίδια χώρα. Γιατί είναι ένα θέμα που βεβαίως και μας απασχολεί πολύ και είναι σοβαρό, αλλά είναι επίσης και ένα θέμα όπου συχνά αμφισβητούνται τα δεδομένα. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την επιδείνωση όσον αφορά τη ισότητα, μάλλον ανισότητα. Έπειτα θέλω να σας ρωτήσω και για την γεωγραφική κατανομή των fake news, εν μάλιστα των ευρωεκλογών. Είναι από τα πράγματα που παρατηρείτε, που εκφράζεται ποσοτικά αυτές οι ψευδείς ειδήσει. Διαπιστώνετε το φαινόμενο να επιδεινώνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γι' αυτό μου αρέσει να έρχομαι εδώ, γιατί πάντα τα θέματα που μου θέτετε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Όσον αφορά τις ανισότητες πρώτα απ' όλα. Εξαρτάται κατά πολύ από την ε, σωστή ερώτηση που βάζουν οι πολιτικοί, τι θέλουν να ξέρουν. Γιατί αν δούμε το Ευρώπη 2020, ο στόχος ήταν να βγει ο κόσμος από την φτώχεια. Βέβαια η κρίση έφερε πολύ περισσότερο το θέμα των ανισοτήτων. Και γίνονται συζητήσεις που δεν είναι καθαρά θέμα στατιστικών δεδομένων. Έχει να κάνει με τους πιο πλούσιους 20 με τους λιγότερο πλούσιους 20, διακρίνονται ομάδες, όπως για παράδειγμα οι νέοι. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Έχουμε δεδομένα, αλλά το θέμα είναι αυτά τα δεδομένα, την πληροφορία, πώς μπορούμε να την ε, διαδώσουμε. Εξαρτάται από την οπτική γωνία του κάθε πολιτικού, του κάθε του καθενός που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό και ο κανονισμός για τα κοινωνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Προσπαθούμε να δούμε το θέμα του εισοδήματος και το θέμα του πλούτου, διαμορφώνοντας τα ασφαλιστικά δεδομένα του μέλλοντος. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται πληρέστερα στοιχεία. Όσον αφορά τώρα τις ψευδείς ειδήσει. Πολύ σύντομα. Δεν μπορούμε απλώς να παρατηρούμε το τι συμβαίνει. Γι' αυτό, μαζί με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δικιά μας άποψη είναι ότι η Eurostat πρέπει να αποτελεί σημείο αναφορά υψηλής ποιότητας με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Συνεπώς, προσπαθούμε να ε, εκτεθούμε στα μέσα ενημέρωσης και οποιοδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μας να μπορεί να το κάνει για να ελέγξει. Συνεργαζόμαστε με τις αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διάφορες ε, χώρες μέλη, γιατί όπως καταλαβαίνετε η γλώσσα παίζει ρόλο εδώ. Όλοι θέλουν να χρησιμοποιούν τη δικιά τους τη γλώσσα, δεν θέλουν να πηγαίνουν ε, στη Eurostat και να τα βρίσκουν μόνο στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά. Οπότε προσπαθούμε έτσι να δημιουργήσουμε εταιρικές σχέσεις, συνεργάτες και συνεργαζόμαστε και με το δικό σας γραφείο ερευνών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε τι προτιμούν, τι είναι αυτό που του χρειάζεται περισσότερο από τα δικά μας τα δεδομένα. Πάντως τα δικά μας τα δεδομένα θέλουμε να τα προβάλλουμε και να είναι εύχριστα, να χρησιμοποιούνται όσο γίνεται από περισσότερο κόσμο. Δεν είμαστε βέβαια οι κυβερνήσει ή η κομισιόν που παρακολουθεί το τι γίνεται, Εμεί τα δεδομένα δίνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ κυρία Κοτσέβα για την πολύ καλή και ενδιαφέρουσα αυτή η επισκόπηση τη τρέχουσα ε, κατάσταση και τη πρόοδου των εργασιών σα και σα εύχομαι κάθε επιτυχία στο πολύ απαιτητικό αυτό καθήκον που έχετε αναλάβει να φέρετε την Ευρώπη πιο κοντά στου πολίτε και νομίζω ότι όπω μα τα περιγράφετε τα πράγματα, ε, η έμφαση στην ιστοσελίδα, στα δεδομένα, με ποια μορφή είναι διαθέσιμη του Ευρωπαίου πολίτε, είναι κάτι ε, πολύ θετικό ε, και σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ελπίζω να σας καλωσορίσουμε ξανά στο Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία. Σας ευχαριστώ. Και εγώ το περιμένω και χρειάζομαι την υποστήριξή σας γιατί έχουμε ένα στενόχρονο διάγραμμα μπροστά μας. Ja, liebe ähm, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι λέω, περνάμε στο σημείο 6 της Μερίσιας Διάταξης Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019. Έχουμε τον εισηγητή μας εδώ, τον Τόμ Βάντε Καντέλα Ρε. Μάλλον δεν τον έχουμε είναι όμως εδώ ο Φάρμπερ, ο Μάρκους Φάρμπερ, Φέρμπερ, που θα τον αντικαταστήσει. Πέντε λεπτά νομίζω ότι του φτάνουν. Έχουμε και 322 τροπολογίες μέχρι στιγμής. Και υπάρχουν και από τη Ρέγκη, τη ΦΑΜ και την γνώμο γνωμοδοτήσεις, όχι από την budget που είναι και η Συνδεδεμένη Επιτροπή. Ο κύριος Φέρμπερ έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Για να μας κάνει μια εισαγωγική παρουσίαση. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Α, αυτό είναι το μικρόφωνο, το σωστό, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο Τόμ δεν μπορεί να είναι εδώ και εκφράσει την ε, λύπη του, αλλά είναι άρρωστος και του ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, βέβαια. Η ασθένειά του πάντω είναι ο λόγο που δεν μπορούσε να είναι εδώ, αλλά μου έχει δώσει ένα μικρό σημείωμα που θα σα το αναγνώσω. Ω εισηγητή έκονα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2019, ο Τόμ ευχαριστεί πρώτα απ' όλα όλε και όλου εσά που συντάξατε επικοδομητικέ τροπολογίες. Η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει πολιτικό χαρακτήρα λέω και εγώ τώρα ε, δεν μας εκπλήσει αυτό και συνεχίζουμε τα λόγια του εισηγητή. Είναι καλό να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Και αυτό έχουμε κάνει και σε διάφορες συναντήσεις και οδών εισηγητών. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες είχαμε επικοδομητικές συναντήσεις. Ο Τόμ ε, επίσης εκφράζει την ε, ευχαριστήσεις του στους και όλους εισηγητές για το επικαιδημοτικό πνεύμα που επέδειξαν στις συζητήσεις ή τη σκέψη για την ανάπτυξη κομισιών θέτει μακροοικονομικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθοδήγηση που έχει τρεις άξονες διασυνδεδεμένους. Πρώτον, δημοσιονομική εξυγίαση, δεύτερον, επενδύσεις και τρίτον, δομικές μεταρρυθμίσεις. Εμείς τώρα πρέπει να αναλύσουμε αυτό το ενάρετο τρίγωνο, αν θέλετε, για να δούμε τις προτεραιότητες αυτές, να, θεωρήσουμε, να πούμε τι είναι ε, τα απαραίτητα για μας μέτρα πρέπει να ληφθούν από Κομισιόν και Σύμβουλο. Τόμ θέλει να εκφράσει την άποψη ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική προτεραιότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γέραση του πληθυσμού και το πώς ε, θα επηρεάσει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ε, και το κράτος πρόνοιας. Ε, ο Τόμ λοιπόν στο σχέδιο έκθεσής του κάνει λόγο για τη γέραση του πληθυσμού θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτό τον άλλο τρίγωνο και στις σχετικές μεταρρυθμίσεις και θεωρεί ότι υπάρχει ευρία στήριξη από τι πολιτικέ ομάδε. Στου δώσαμε έμφαση και στην ανάγκη να έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, δυναμικό ε, εργατικό δυναμικό. Η επιμόρφωση, η διαβίου θα είναι το νέο πρότυπο, ο νέος κανόνας. Πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας. Επίσης, σχέδιο σε σχέση με το σχέδιο έκθεση. Μεγαλύτερη έμφαση στι επενδύσει, στη γενειακή δικαιοσύνη. Σημαίνει και προοδευτικέ ε, επενδύσει στραμμένε προ το μέλλον. Δημόσιε επενδύσεις, επενδύσει, δεξιότητε, έρευνα ανάπτυξη, υποδομέ. Κυρίω όμω στην καινοτομία, στον στην αυτοματοποίηση, στην ψηφιοποίηση. Αύριο θα ψηφίσουμε την έκθεση ώστε να στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σαφές μήνυμα προς Κομισιόν και Συμβούλιο. Στόχο είναι να μην έχουμε χωριστέ ψηφοφορίες στην έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να πάει πάρα πολύ καλά η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ Μάρκους που εξπροσώπησε τον εισηγητή μας. Ο Πέτρος Σίβα Περέρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχηθώ καλή τύχη. Για την... Ε, ελπίζω ο συνάδελφος να συνέλθει σύντομα και να είναι μαζί μας γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό το ντοσχέ. συζητούμε τους προσανατολισμούς της δημοσιονομικής πολιτικής και πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και ως όδης εισηγητής θέλω να επιβεβαιώσω ότι ήταν πολύ πρόσφορη η όλη δουλειά που έγινε στις συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών. Είναι αλήθεια ότι πολλές τροπολογίες υποβλήθηκαν και μάλιστα Πολλέ τροπολογίε θα πει και πολλή δουλειά, έτσι. Έχουμε δουλέψει σκληρά. Και αν οι τροπολογίες αυτές είναι το αποτέλεσμα αντικρουόμενων πολιτικών απόψεων, και αυτό είναι ο λόγο που είναι πολλέ, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. Όμω ο εισηγητή ήταν αρκετά ε, διαλλακτικό ώστε να λάβει υπόψη τις βασικές μας μπέριμνε. Έχουμε αναδιοργανώσει και αναδιαρθρώσει τελείω την έκθεση σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Τώρα είναι πολύ πιο καλά εξισορροπημένη η όλη προσέγγιση και πιστεύω Πιστεύω ότι η έκθεση σε σχέση με τις τροπολογίες και τις συμβαστικές που έχουν ε, συζητηθεί θα μπορέσει να επιτρέψει να προκύψει μια ισχυρή θέση στο Κοινοβουλίο σε αυτή την ε, κρίσιμη στιγμή για την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Κατά την άποψή μας το πιο σημαντικό είναι να έχουμε κάποια απάντηση στην ε, οικονομική ύφεση, την οικονομική αυτή αργοπορία που παρατηρούμε και στα δημοσιονομικά και στα οικονομικά μας φαίνεται αυτό. Είναι σημαντικό ε, να πούμε ότι τώρα αναγνωρίζεται πλέον το επενδυτικό χάσμα στην Ευρωζώνη και η ανάγκη να υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτό μέσω επενδύσεων κοινών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, Τώρα στην έκθεση υπάρχει σαφής στήριξη προς τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναγκάσει τα κράτη-μέλη με μεγάλο πλεόνασμα στο αγαθάριστο εισόδημά τους να κάνουν κάτι για να ενισχυθεί η ζήτηση και να υπάρξει περισσότερη κίνηση στις επενδύσεις. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να υπάρξει μια υγιής δημοσιονομική πολιτική και τέτοιες επενδύσεις ε, θέλουμε στον τομέα τον κοινωνικό και σε άλλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εκτελεστούν το λόγο της ε, το στόχο της συμμετοχής όλων μάλλον τώρα λαμβάνεται υπόψη οπότε πιστεύω ότι έχουμε ε, αρκετά δεδομένα για να πετύχουμε μια ευρεία συνένεση στο, στο Κοινοβούλιο στην εξέταση του όλου θέματος. Ευχαριστούμε Πέντρο, Σίλβα, Περέιρα. Δεν είναι κανείς εδώ από τους συντηρητικούς, τα απ' την άλλη. Πράσινη, κανείς. Δεν βλέπω κανέναν εδώ, ούτε και από την ΚΟΕ. NGL. Ούτε το ENF εκπροσωπείται. Άρα τελευταίος και καλύτερος ο συνάδελφος Μάρκο Βάλλη από την EFTD. Ευχαριστώ Πέτερ. Ε, πολύ γρήγορα. Κάθε φορά επί τη διαδικασία του εξαμήνου υπάρχουν διαφορετικέ πολιτικέ θέσει. Γιατί είναι δύσκολο να καταρτήσουμε μια κοινή οικονομική πολιτική, φυσικά. Ε, γι' αυτό οι ειδικέ εκθέσει που βλέπουμε κάθε χρόνο ε, συνήθως ε, είναι εκθέσεις που συνοδεύονται και πάρα πολλές δικές μας τροπολογίες. Δεν συμμεριζόμαστε όπως γνωρίζετε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια στρατηγική που σκοπό έχει μόνο να συγκρατεί τις δαπάνες με μέτρα λιτότητας και μεταρρυθμίσεις που πολύ συχνά ε, χτυπάνε και υποβαθμίζουν τους μισθούς, ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θέλουν να κάνουν πιο ανταγωνιστική την Νότια Ευρώπη, όμω είναι μεταρρυθμίσει κοινωνικά άδικε και μη βιώσιμε και από κοινωνική σκοπιά και οικονομική. Και ω προ την κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων, που πολλέ φορέ θα μπορούσαν να αποφευθούν. Γιατί πρόκειται για υποθέσει πολύ λεπτές που πρέπει να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τώρα τι προσπάθειες που απαιτούνται, διαρκώ απαιτούνται προσπάθειε στι χώρε με υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα και άλλε δυσκολίε και δεν γίνεται κάτι για το άλλο σκέλος του προβλήματος στην Ευρωζώνη, που είναι το πλεόνασμα στο τρέχοντες λογαριασμού κάποιων κατώμελων στο ΑΕΠ όπως η Ολλανδία εδώ και πολλά χρόνια, που έχει υπερβολικά πλεονάσματα επί χρόνια επαναλαμβάνουμε ότι από το όριο των 6% και μετά θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική διαδικασία και για αυτές τις χώρες. Θα έπρεπε να υπάρχει ε, Ε, μια ε, πολιτική σωστά εξορπημένη, όχι μόνο ιδιαίτερη επιθετικότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις περιπτώσεις των ε, δημοσιονομικών ελλημάτων και το άλλο σκέλος είναι πολύ σοβαρό για την υγεία της Ευρωζώνης. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι στην έκθεση αυτή αυτό που δεν έχει γίνει είναι ότι το σύμφωνο, δεν έχει πιστεί ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξη έχει εφαρμοστεί κάθε φορά ανάλογα με το χρώμα της κυβέρνηση που κυβερνά την κάθε χώρα εντό τη Ευρωζώνη. Αρκεί να σκεφτούμε τα τελευταία γεγονότα σε σχέση με το γαλλικό έλλειμμα και τις παραμέτρους του Μάστριφτ. Δεν ελήφθη υπόψη, όπως θα έπρεπε, το υπερβολικό έλλειμμα της Ιταλίας και κάποιες άλλες υπερβάσεις Οι τεχνικές ενδείξεις λοιπόν και οι επισημάνσεις που έχουν γίνει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο θα έπρεπε να ληφθούν διαφορετικά υπόψη. Από δική μας πλευράς λοιπόν καλό θα ήταν στο κείμενο κάτι να αναφέρεται, μια πρόταση για δημοσιονομικές μεταφορές ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες που υπάρχουν, ε, τα χάσματα και τα κενά που υπάρχουν στην Ευρωζώνη. Δεν μπορεί οι χώρε με τους τρέχοντες λογαριασμούς με τεράστια πλεονάσματα να μην συνεισφέρουν καθόλου στην επίλυση των διαφορετικών προβλημάτων των επενδύσεων στο Νότο. Και για τις επενδύσεις αυτές θα πρέπει να οριστεί και ένας στόχος για να γίνουν ε, μαζικές δημόσιες επενδύσεις και να μπορέσουν οι χώρες αυτές να ξεφύγουν λίγο από την ε, πορεία αυτή του φαύλου κύκλου. Ε, Δυστυχώ πολλέ από τι προτάσει μα δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο, αλλά αυτό δεν θα μα κάνει να μετατοπιστούμε από τι απόψει μα. Ευχαριστώ και τον Μάρκο Υπάρχει κάποιο που θα ήθελε το λόγο στο πλαίσιο τη έντυπη κάτι Όχι. Κύριο Φέρμπερ, θέλει να πει κάτι εκ μέρους του εισηγητή καταληκτικά. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που συμμετείχαν και στη σημερινή συζήτηση, αλλά και στις πολύ επικοδομικές συναντήσεις των σκιωδών και αύριο ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ισχυρή τοποθέτηση ως κοινοβούλιο, αρχικά ως έκον και εν συνεχεία ως κοινοβούλιο, προς την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Φέρμπερ. Νομίζω ότι καλύπτονται και 322 τροπολογίες από τις συμβιβαστικέ που θα ψηφίσουμε αύριο. Και ελπίζοντας ότι θα πάει καλά η αυριανή ψηφοφόρια, θα ψηφίσουμε και στη δεύτερη σύνοδο του Μαρτίου του 2019, οπότε κλείνουμε και αυτό το σημείο της μεσιάς διάταξης και πολύ νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα. Αλλά ο ψηγητής ε, δεν μπορεί να είναι εδώ, το ήξερα από πριν, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε, έχετε όλοι το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. μπορούμε ήδη να ξεκινήσουμε από τις 6 παρα 25 και όχι στις 6 όπως προβλεπόταν το επόμενο σημείο γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ο συγητής Μιγγέλ Βιέγας της ΓΚΟΕ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Με παρακάλεσε όμως να διαβάσω μία ανακοίνωση εκ μέρους του. Κύριος Βιεγάς. Έγκας λοιπόν μου λέει να σας πω τα εξή. Αυτή η πρόταση είναι μέρος ενός πακέτου προτάσεων για το, από το Μάιο 2013. Η Επιτροπή προτείνει κανόνες λοιπόν για τους ειδικού φόρους που θα καλύπτουν τους ειδικού φόρους για το αλκοόλ. Η οδηγία προηγούμενη, 92-83 θέτει τους κανόνες για τους φόρους αυτούς, για την παραγωγή, την αποθήκευση αλλά και την διακίνηση τέτοιων προϊόντων μεταξύ των χωρών μελών. Στόχο τη οδηγία αυτή είναι να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών αυτών, διασφαλίζοντα συγχρόνω όμω ότι οι φόροι συλλέγονται από τη χώρα μέλο που πρέπει. Η οδηγία λοιπόν έχει τροποποιηθεί πολλές φορές μέχρι τώρα. Η οδηγία επίσης περιλαμβάνει διάφορες αναφορές σε νομοθεσία που πρέπει συγχρόνως να ενημερωθεί. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την επαναδιατύπωση της οδηγίας 2008-118 ΕΚ ε ο εισηγητή λοιπόν, ο κύριος Μιγγέλ Βιέγκα, λέει ότι συμφωνεί με το πνεύμα και με το περιεχόμενο τη πρόταση αυτή. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα, θα προχωρήσουμε προτείνει με απλοποιημένη διαδικασία και δηλαδή να ψηφίσουμε την έκθεση χωρίς τροπολογίες. Αυτή είναι η πρόταση του εισηγητή. Να πάμε στην απλοποιημένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες. Θα δώσω το λόγο στον σκιώδη των σοσιαλιστών Όλε λούπκισον. αλλά, αλλά συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη. ξέχασα σε αυτό το σημείο ότι εδώ ο Μάρκος πρέπει να πάρει το λόγο. Ο Μάρκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, δυστυχώς θα αλλάξουν τα πράγματα μετά τις ε, εκλογές ίσως, πάντως προς το παρόν το ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα σε αυτό το σώμα. Οπότε ναι, εμείς μιλάμε πρώτα. Λοιπόν, η πρόταση αυτή θέτει τις διευθετήσεις για τους ειδικού φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς επίσης και τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Η οδηγία έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή, την αποθήκευση και τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικού φόρου κατανάλωση μεταξύ των κρατών μελών. Ο κύριο στόχο τη οδηγία είναι να καταστεί δυνατή ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι τα κράτη-μέλη εισπράττουν εν τέλει την ορθή φορολογική οφειλεί. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τεχνικό μέτρο, ε, δεν είναι επίμαχο πολιτικά και δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει τόση πολλή δουλειά και λίγο χρόνο, γι' αυτό εμείς το ΕΛΚ συμφωνούμε με τη θέση του εισηγητή να προχωρήσουμε με την απλοποιημένη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μάρκος Φέρμπερ για το ΕΛΚΑ και τώρα για τους Εσλιστές και Δημοκράτες. Όλοι λούντξαν Σκιώδης. Ευχαριστώ. Είναι θετικό που μπορούμε και συζητάμε για την απόφαση αυτή να έχουμε μια απλοποιημένη διαδικασία και να αποφύγουμε οποιαδήποτε ε, φοροδιαφυγή. Αυτό που θέλουμε είναι να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η διοικητική διαδικασία και οι δηλώσεις των τελωνιακών αρχών όσον αφορά τα προϊόντα που υποβάλλονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο της φόρο αποφυγής και της φόρο διαφυγής όσον αφορά τα προϊόντα αυτά που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γι' αυτό και συμφωνήσαμε με τον εισηγητή τον κύριο Βέγκας και θέλουμε και εμείς να εγκρίνουμε με την απλοποιημένη διαδικασία της ε, τροπολογίας και τις αλλαγές σε αυτό το κείμενο. Ευχαριστούμε επόμενος δεν είναι εδώ. Απ' την άλλη κανείς. Σελσκάτο από τους πρασίνους δεν είναι εδώ. Οπότε ερχόμαστε στη διαδικασία Κατσδιάη. Συνεπώς, έχω να κάνω την εξής πρόταση, αφού δεν υπάρχει κανείς. Κανονικά, κανονικά, πρέπει να ρωτήσω αν έχει κάποιο αντίρρηση από την αίθουσα. Και αν δεν υπάρξουν 7 που έχουν αντίρρηση, τότε πρέπει να δεχτούμε την πρόταση αυτή για απλοποιημένη διαδικασία. Δεν είμαστε καν 7 στην αίθουσα όμως. Οπότε Έχω την εξής πρόταση για να είναι σαφές ότι τυπικά, νομικά, αυτό που κάνουμε στέκει. Λοιπόν, ολόκληρη η Επιτροπή, οι συνάδελφοι που είναι εδώ και όσοι δεν είναι εδώ, αν έχουν αντίρρηση να το πούνε στην γραμματεία μέχρι τις 10 το πρωί αύριο πρέπει να υπάρχει γραπτή αντίρρηση, ώστε νομικά να είμαστε καλυμμένοι. Έτσι. Αν δεν υπάρξουν 7 ή παραπάνω τέτοιες ενστάσεις μέχρι αύριο το πρωί στις 10, τότε θα συνεχίσουμε και θα ακολουθήσουμε την προτινόμενη απλοποιημένη διαδικασία όπως προτείνει ο κύριος Βέγας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτά για σήμερα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αύριο συνεχίζουμε από τις 9 το πρωί με την ανταλλαγή απόψεων με τον ε, κύριο Hans Hocherforst, πρόεδρο του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τον Μισελ Πράντα, πρόεδρο των διαχειριστών τόνο του Ιδρύματος ΔΠΧΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έληξε η σημερινή συνεδρίαση.